και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είστε διατεθειμένοι να μας υποστηρίξετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξεχθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο σημερινή σε διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Ολένια η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής θάλασσας και ο ρόλος των μακροπεριφερειών στη μελλοντική πολιτική συνοχής. Τον λόγο έχει ο εισηγητής για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές για το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν, χάρη στο οποίο έχουμε καταφέρει να συντάξουμε την έκθεση αυτή. Αναφέρεται στις μακροπεριφέρειες, στην στρατηγική για την περιοχή της Βαλτικής, και τη σημασία αυτής της πολιτικής για την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφερόμαστε στις μεταφορές στη γεωργία, έρευνα και ανάπτυξη. Το 2004 αρχίσαμε να μιλάμε για το θέμα αυτό. 8 από τις 9 χώρες της Βαλτικής ήταν τότε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολιτικέ μεταφορέ εδώ αναφέρονται ω προτεραιότητε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί θα πρέπει να συνενώσουμε τι δυνατότητέ μα και τι υποδομέ μα για να επιτύχουμε του στόχου αυτού. Μιλάμε για μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση στι μακροπεριφέρειε αυτέ. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, παραδείγματο χάρη, την ρήπανση, είναι απαραίτητο να μην το κάνουμε αυτό με ω κράτη-μέλη. Θα πρέπει να προωθήσουμε τη συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών σε μια μακροπεριφέρεια γιατί αυτό είναι και μοχλός για την οικονομική ανάπτυξη και μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τις ικανότητες των ανθρώπων, τα ταλέντα τους που ζουν στην περιοχή της Βαλτικής. Αν το πετύχουμε αυτό, τότε θα συμβάλλουμε και στην ανάπτυξη του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η περιοχή της Βαλτικής είναι πρωταρχική σημασίας για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δημιουργήσουμε πλούτο προς το όφελος όλων των λαών της περιοχής. Και αυτό θα γίνει κυρίως μέσα από την παιδεία. Θέλουμε να προωθήσουμε την κοινωνία των πολιτών επίση γιατί αυτό. και είναι και η βάση ενό δημοκρατικού συστήματο. Αν το πετύχουμε αυτό, τότε θα υπάρξει όλο και μεγαλύτερη ενσωμάτωση και ολοκλήρωση μεταξύ των χωρών τη περιοχή. Αυτά τα αποτελέσματα όμω δεν μπορούν να επιτευχθούν εάν δεν ανυψώσουμε και το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων τη περιοχή. Αυτό μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Είναι μια τεράστια πρόκληση ενώπιών μας. Έχουμε πιλωτικά προγράμματα για τη δημιουργία της μακροπεριφέρειας αυτή στην περιοχή της Βαλτικής. Και αυτό σημαίνει μια σειρά από σχέδια και πρωτοβουλίες για την περιοχή της Βαλτικής και κατά την άποψή μου θα πρέπει να θα πάντα ότι κάποια συγκεκριμένα μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν κάτι το οποίο απαιτεί και τη χρηματοδότηση αυτών των πρωτοβουλειών στην επόμενη περίοδο δημοσιονομικού σχεδιασμού. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθηθεί στο να, να κατατήσει μια βάση βελτίστων πρακτικών η οποία θα είναι χρήσιμη το μέλλον. Θέλουμε λοιπόν όλα αυτά τα προγράμματα να είναι αποτελεσματικού χαρακτήρα και φυσικά να μεταλαμβανευτεί η εμπειρία μας και σε άλλες μακροπεριφέρειες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητούμε από την Κομισιό λοιπόν να υποστηρίξει και να προστατεύσει την ιδέα αυτή. Όταν φτάσουμε λοιπόν στην ενδιάμεση αναθεώρηση αυτή τη αδίκη, αυτά τα οποία θα έχουμε επιτύχει εμεί, θα είναι το σημείο αναφοράς για άλλα παρόμοια προγράμματα στο μέλλον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση. Και επίση θα πρέπει να δώσουμε τι απαραίτητε απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία έχουμε ενώπιόν μας. Θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν αυτέ οι πρωτοβουλίε από την πολιτική συνοχή ή να υπάρχει συγκεκριμένη μνήμα στον προπολογισμό. Εγώ χαίρομαι που η αρχή τη μακροπεριφέρεια άρχισε να αναπτύσσεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα. Μπορούμε μέσω αυτή να προωθήσουμε την εδαφική συνοχή και αυτό είναι ένα από του καλύτερου τρόπου να προωθήσουμε τι οδηγέ και ιδρυτικέ ιδέε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αναπτύξουμε περιοχέ και περιφέρειες που έχουν κοινά συμφέροντα και τη δυνατότητα συνεργασία. Η περιοχή τη Βαλτική είναι φάρο προ την κατεύθυνση αυτή μπορούμε να αποδείξουμε το σύστημα αυτό λειτουργεί και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση λειτουργεί. Ευχαριστώ. Kelly, Zapata, Boris, Kalinowski, Lumen, Senalova, Tabaji, Kursky. Mr. Kelly, one minute or less. Come on, Tron. Those Tommy Vavor on Strategia Πράγματι πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση που δεν αφορά μόνο το βόρειο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπλέκεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν χρειάζονται επιπλέον χρήματα, επιπλέον κονδύλια, δεν θα κοστίσει δημοσιονομικά, δεν απαιτείται νέο νομικό πλαίσιο, δεν απαιτείται η δημιουργία περιττέρω θεσμικών οργάνων. Απλά θα πρέπει να λύσουμε σε επίπεδο περιφερειακό κάποια προβλήματα κοινά σχετικά με το περιβάλλον που ενδιαφέρουν τις κοινωνίες της περιοχής αυτής. Η στρατηγική αυτή λοιπόν νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη και θα πρέπει να χρησιμεύσει σαν παράδειγμα και για άλλες περιοχές. Ζασάντα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είμαι πεπισμένος ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής θα οδηγήσει σε ε, περισσότερο αηφόρο μορφές ανάπτυξης. Θα πρέπει όμως παρόλα αυτά να ελέγχουμε τις διαδικασίες αυτές. Νομίζω ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή αυτή είναι να δημιουργήσει ένα ουσιαστικό δίκτυο μεταφορών είτε θαλασσίων, είτε εσωτερικών υδάτινων πόρων, είτε οδικών. Και γι' αυτό ακριβώς η τροπολογία μου σχετικά με την δημιουργία δικτύων ε, και διαδρόμων οδικών έχει ε, συμπεριληφθεί νομίζω ότι υπάρχει η δυνατότητα να συνδέσουμε με σωστό τρόπο το σύνολο των περιχών αυτής της περιφέρειας. Να βελτιώσουμε λοιπόν τις υποδομές, βελτιώνοντας την επικοινωνία ανάμεσα στις πόλεις και τους πολίτες φυσικά. Έχει τεράστια σημασία λοιπόν το πρόγραμμα αυτό, όχι μόνο οικονομική αλλά και πολιτιστική και ιστορική. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Ολένιτσακ για την εξαιρετική της έκθεση. Η πολιτική συνοχή είναι μια καινούργια πρόκληση. Οι μακροπεριφέρειες είναι μια ενδιαφέρουσα έννοια. Αναφέρονται στη Μεσόγειο, στη Βαλτική και εδώ μιλήσαμε για ένα μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή του θέματος όχι μόνο τη Βαλτική αλλά και τη Μεσόγειο. Οι θάλασσες αυτές πρέπει να ενωθούν μεταφορικώς, να βρεθεί ένας διάδρομος ώστε να υπάρξει αμοιβαία ανάπτυξη. Ξέρω ότι ακόμα γίνονται διαπραγματεύσεις για τις διασυνδέσεις ε, οδικός ή σιδηροδρομικός και είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό αν θέλουμε να υπάρξει πράγματι συνοχή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Επιτροπή Μεταφορών επισκέφθηκε την Εστονία και τη Λετωνία και συζήτησε μαζί με τους αρμοδίους των χωρών αυτών την κατάσταση μεταφορών. Δεν μιλάμε μόναχα για διασύνδεση προς το Ανατολικό α, μέρος Ευρώπης, αλλά και υπέρβαση των σημείων συμφόρησης που παρατηρούνται στις μεταφορές στην περιοχή αυτή. Υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τη διασύνδεση των χωρών αυτών και γι' αυτό θα πρέπει να υπογραμμίσουμε και το να έχουμε αυτόν τον διάδρομο ο οποίος συνδέει την Βαλτική και τη Μεσόγειο από την Αδριατική. Νομίζουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούμε να έχουμε ένα σημαντικό θετικό αντίκτυπο για όλες τις χώρες της περιοχής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ολενίτσακ για την έκθεσή του η στρατηγική για την ανάπτυξη της μακροπεριφέρειας της Βαλτικής είναι μια ιδιαίτερα επιτυχή στρατηγική για εμά. οι οποίοι ζούμε στην περιοχή αυτή θα θέλαμε να δούμε να δημιουργηθεί η περιοχή γιατί και εμείς επιζητούμε κάτι αντίστοιχο για την περιοχή του Δούναβη. Είναι σημαντικό λοιπόν τα παραδείγματα αυτά να ευδοκιμήσουν. Δεν πρέπει να καθορίσουμε υπερβολικά πολλές προτεραιότητες. Θα πρέπει να έχουμε τους δύο-τρεις κύριους στόχους που είναι αυτοί οι οποίοι θα φέρουν κοντά τις ε, χώρες τις όμορες του Δούναβη, όπως και για τις ε, χώρες της Βαλτικής. Είναι κυρίως τα θέματα μεταφορών, όπως η πλοημότητα του Δούναβη και η εξασφάλιση της βιοποικιλότητας και της ποιότητας των υδάτων του Δούναβη και επίσης και η ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων. Εγώ πιστεύω ότι η επερχόμενη Ουγγρική Προεδρία το 2011 θα θεωρήσει αυτή τη διαδικασία σαν μια προτεραιότητα και είμαι υπερήφανος διαπιστώνω ότι ο κ. Σεφκοβιτς ως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να παίξει και αυτός ένα ρόλο για να αναδυθεί αυτή η μικρο η μακροπεριφέρεια στην περιοχή, στην περιοχή του Δούναβη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι από το Κτάνσκ στην Βαλτική και φυσικά υποστήριζω αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα της ανάπτυξης μιας μακροπεριφέρειας. Έχω μονάχα δύο επιφυλάξεις. Εγώ θέλω να υπάρξει μια πιο εύρωστη πρωτοβουλία αυτό απαιτεί χρήματα, Επομένω πρέπει να έχουμε του ίδιου πόρου στην ίδια χρηματοδότηση. Χωρί αυτά απλώ μιλάμε στον αέρα ή στο νερό. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώ θα έχουμε και περισσότερη χρηματοδότηση για αυτήν την στρατηγική, Αλλιώ θα υποχρεθούμε να κάνουμε περικοπέ σε άλλα προγράμματα για να μπορούν αυτά τα σχέδια να ευδοκιμήσουν. Αυτό θα είναι ολέθριο. Μια δεύτερη επιφύλαξη. <clears throat> Δυστυχώ η Βαλτική είναι ακόμα μία από τι πιο ρηπασμένε θάλασσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ και το North Stream ο αγωγός αυτός παίζει κάποιο ρόλο. Θα πρέπει να μειώσουμε την εξάρτησή μας από την παροχή φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μια συνεκτική στρατηγική για τα θέματα αυτά. Είδαμε να υπάρχει καταρχήν το όχι και μετά το ναι για το North Stream. Καλή για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Λένιτσακ. Πρόκειται για μια καινοτομία, όχι μόνο για την περιοχή αυτή, αλλά για το βορρά της Ευρώπης γενικότερα και εφόσον επιτύχει ίσως να υπάρξουν και περαιτέρω τέτοιου είδους συνεργασίες. Θέλουμε εμείς να ανοίξουμε τις ευκαιρίες και να διασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες για όλους. Θέλουμε να καλυφθούν οι καθυστερήσεις στην ανάπτυξη σε ορισμένες περιοχές και θέλουμε να καθοδηγήσουμε σωστά την οικονομική ανάπτυξη των χωρών που συνορεύουν με τη Βαλτική θάλασσα. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι μια σωστή συνεργασία και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών διμερών σχέσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η στρατηγική της Βαλτικής στην μακροπεριφέρεια αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι έχουμε μια ενσωματωμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη όλες τις δυνατότητες και τις προκλήσεις στην περιοχή και είναι και ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Η στρατηγική αυτή λοιπόν μπορεί να αποτελέσει ένα υπόδειγμα για μελλοντικές εφαρμογές στρατηγικών σε άλλες περιοχές τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ περιλαμβάνεται και αυτή που αφορά το Δούναβι. Τα ευρωπαϊκά σχέδια μπορούν να έχουν ένα σημαντικό ρόλο για τις περιοχές αυτές και να παίξουν τον πρέποντα ρόλο. Όλα αυτά είναι πολύ απαραίτητο να γίνουν με τη συμμετοχή των κρατών μελών, με όλα τα κονδύλια τα οποία έχουν δοθεί για αυτά τα προγράμματα. Και πρέπει να υπογραμμίσω περαιτέρω το γεγονό ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τι ιδιαιτερότητε αυτών των περιφερειών, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει και σε μια καλύτερη χρησιμοποίηση των κοινωνικών ταμείων και δημιουργία τοπικής προσθέμενης αξίας. Uh, για μια ακόμη φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λέσνιτσακ για την έκθεσή του, όπως επίσης και για την αιμονή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Βαλτική περιοχή. Αυτή η νέα περιοχή ελέγχει ουσιαστικά, περνάει από τεστ τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμεθα και εξετάζει τη συνέχεια που δίδουμε στις αποφάσεις που λαμβάνουμε. Είναι σαφές ότι η ουσιαστική συμμετοχή όλων των εμπλικωμένων περιοχών ε, θα είναι καθοριστική. Για πρώτη φορά έχουμε προετοιμάσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για μια σειρά κρατών που αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις και που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις, ευκαι... από ίδιες ευκαιρίες. Το κάνουμε αυτό λαμβάνοντας υπόψη τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μάλλον κάθε χώρας και δημιουργούμε νέες μεθόδους συνεργασίας με τις κυβερνήσεις. Για πρώτη φορά προσπαθούμε να συνδυάσουμε τις δυνατότητες που έχουν οι διάφορες χώρες συνδυάζοντας ταυτόχρονα και τις, ε, και τις διάφορες πολιτικές και τα διάφορα προγράμματα που έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε την περιοχή μακροοικονομικά. Περιβάλλον, θέματα ασφαλείας, θέματα ενέργειας, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα και εκεί η αποτελεσματικότητά μας θα μεγιστοποιηθεί από τα νέα αυτά. Νομίζω ότι η αντιμετώπιση αυτή έχει ήδη αποδειχθεί στο παρελθόν επιτυχής. Ακριβώς έχουν υπάρξει προγράμματα που αφορούν πολλές από αυτές τις χώρες που έχουν χρηματοδοτηθεί από τα Ταμεία Συνοχής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να διατηρήσει την όθηση την οποία έχουμε πετύχει μέχρι τώρα η συνάντηση στο Καλίνιγκρατ στις 14 και 15 ε, Οκτωβρίου θα μας δώσει την δυνατότητα να διαπιστώσουμε τα αποτελέσματα της πολιτικής μέχρι σήμερα και να δούμε ποιες είναι οι μελλοντικές ανάγκες και πώς θα μπορέσουμε να αναζωογονήσουμε επίσης και το περιβάλλον στην περιοχή αυτή βελτιώνοντας την ποιότητα των υδάτων της Βαλτικής θάλασσας που είναι ένα σημαντικό θέμα. Υπάρχουν ε, πολλά υποσχόμενα προγράμματα τα οποία γίνονται απικείμενο επεξεργασίας και σε επίπεδο οδικών μεταφορών και κάτι το οποίο θα επιτρέψει φυσικά την μεγαλύτερη και καλύτερη ολοκλήρωση της περιοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η μακροπεριφερειακή αντιμετώπιση της συγκεκριμένης περιοχής θα προσφέρει προστιθέμενη αξία νομίζω και σε επίπεδο μεθοδολογικό για άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό θα μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε και στην περίπτωση του Δούναβιτ που είναι σε επίπεδο προπαρασκευής. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει τέτοιου είδους προγράμματα να συγγράφονται στην Τσεχία, στην Σλοβακία συγγνώμη, και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει κατανόηση μεταξύ μας για τις ανάγκες της περιοχής αυτής. Για το αν θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις θα δούμε. Αυτό θα εξαρτηθεί από την επιτυχία των δύο πρώτων προσπαθειών και αν μπορούμε να προσθέσουμε κάτι περισσότερο από τις δυνατότητες τις οποίες ήδη έχουμε στην διάθεσή μας. Ελπίζω λοιπόν, κάθε, εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτούς οι οποίοι ξεκινούν την προσπάθεια στα πλαίσια της στρατηγικής ε, ε, αυτής, ε, όπως επίσης και στην επερχόμενη Προεδρία για την περίπτωση του Δούναβη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και Φτάσαμε εσείς στην τελευταία έκθεση της σημερινής βραδινής συνεδρίας, που είναι η έκθεση της κυρίας Κράτσας Τσαγκαροπούλου σχετικά με τη